να τελειώσει η διάσκεψη των Προέδρων, σχεδόν έχει τελειώσει. Πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίε, έχω δει διαδικαστικά. Από την κυρία Φορέντζα πρώτα. Κυρία Φορέντζα, Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν είναι παραδεκτό βάσει του ιστορικού κανονισμού του Κοινοβουλίου αυτά που είπε ο συνάδελφο Μάρκο Φάρμπερ, ότι η Τρόικα θα έπρεπε να εισβάλλει στη Ρώμη και να πάρει στα χέρια του το Υπουργείο των Οικονομικών. Ήθελα να θυμίσω στον συνάδελφο ότι η Ιταλική Δημοκρατία βασίζεται στην αντίσταση κατά τη βία ε, και αυτό προβλέπει και το Σύνταγμά μα. Δεν ε, μπορεί λοιπόν να παραδοθούμε στον επικρατισμό τη Γερμανία. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ε, κοινωνική δικαιοσύνη και κάποια σεβασμό. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε γνώση αυτών των σχολείων και να τα καταδικάσετε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Σημειώνω όσα είπατε. Έχουμε διαδικαστικό και την κυρία Γκαρθία Πέρεθ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τι ε, κυρώσει ε, προς ε, τον συνάδελφο Κόρβιν Μίκε, ο οποίος είχε προσβάλει και θίξει την αξιοπρέπεια των Ευρωπαίων γυναικών. Θέλω να πω ότι μπορεί να του επιστραφούν τα χρήματα, το πρόστιμο δηλαδή, όμως την αξιοπρέπεια δεν μπορεί να του την επιστρέψει, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σέβονται τη γυναική αξιοπρέπεια. Απέναντι λοιπόν σε τέτοιες τοποθετήσεις και τέτοιες παρεμβάσεις, ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να ε, στηρίζει άκαμπτα και στεναρά τα δικαιώματα των ε, γυναικών. Thank you. Ευχαριστώ. Thank you, Madam. The judgment is just made. Ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς θα το μελετήσουμε. Έχουμε και κάτι ακόμα από έναν συνάδελφο. Παρακαλώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύει την ελευθερία του λόγου εδώ μέσα όταν κάνουμε κήρυγμα σε ολόκληρο τον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να τιμωρούμε κάποιον για κάτι το οποίο είπε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό αυτή η απόφαση είναι θρίαμβος για την ελευθερία λόγου και χαίρομαι που ελήφθη. Ευχαριστώ. Ε, και εσείς διαδικαστικό. Κύριε Γκουαλτιέρη, όχι συζήτηση από του θέματος. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ανέγνωσα με πολύ αντισαρέσκεια ε, τις δηλώσεις του πρώτου μας αντιπροέδρου, του κυρίου Φέρμπερ, ο οποίος κάνει λόγο για το πώς θα έπρεπε η, Ρώμη, η Τρόικα να εισβάλλει στη Ρώμη και να πάρει στα χέρια του το Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω ότι κάποιος με ένα τέτοιο θεσμικό λειτουργήμα δεν μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό του να εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι απαράδεκτο. Περιμένουμε Περιμένουμε επίσημη συγγνώμη και να αποσύρει αυτέ τι απαράδεκτες εκφράσει του ο κ. Φέρμπερ. Διότι θα είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστώ με τον ε, ε, αντιπρόεδρό μου τι προσεχή ημέρες. Ευχαριστούμε. Κύριε Φέρμπερ, θέλετε και εσείς το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ρώτησε η γερμανική τηλεόραση τι θα συνέβαινε εάν η Ιταλία πλέον δεν ήταν σε θέση να πληρώσει και εκεί απάντησα ότι αν δεν είναι πλέον σε θέση θα έπρεπε η Τρόικα όπως συνηθίζεται στην Ευρωζώνη ε, μα αφήστε με να το πω Συνάδελφοι Λοιπόν Μόλις τώρα πανηγυρίζαμε που το δικαστήριο επέτρεψε την ελευθερία έκφρασης. Ελπίζω να ισχύει για όλους εδώ μέσα. Η διατύπωση που ακούσατε δεν ήταν η δική μου διατύπωση, ίσως ήταν θέμα μετάφρασης. Εγώ είπα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς έγινε στο παρελθόν. Αν δείτε το πρωτότυπο δεν είναι τόσο άσχημο όσο αυτό που παρουσιάζεται στην Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσαν τα διαδικαστικά. Αδελφοί, νομίζω καλό είναι να το δούνε πρώτα στην αρμόδια επιτροπή το θέμα αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Να Έχω την αδειά σα να περάσουμε στι ε, ψηφοφορίε. Λοιπόν, ποιοι θέλετε να ψηφίσουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Περνάμε στην πρώτη έκθεση, η κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει το ψήφισμα σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.